Bueno. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε. Παρακαλώ καθίστε. Estamos esperando... Περιμένουμε τον κύριο Μπροκ. Αλλά τρέχει ο χρόνος. Σας παρακαλώ καθίστε, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ καθίστε. Ε, vamos a Δεν θα περιμένουμε τον κύριο Μπροκ. Έχει περάσει η ώρα. Όταν φτάσει, έφτασε. Έχουμε αυτή την ακρόαση για, το για την κατάσταση γνώμη του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Έχουμε τον κύριο Αλή Σαχίν, υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Ήταν στις Βρυξέλλες και εξέφρασε την βούλησή του να μιλήσει στην υποεπιτροπή μας. Τον ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία του και δίνω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Υφυπουργό. Παρακαλώ κύριε Υφυπουργέ. Dear chairs αγαπητοί πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ που με δέχεστε και ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας μετά το ε, πραξικόπημα. Θα ήθελα να μιλήσω στα τουρκικά, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε έτοιμοι με τη μετάφραση. Ωραία. Θα ήθελα να πω το εξής καταρχήν. Μετά τις 15 Ιουλίου η Τουρκία ζει μια καινούρια, ένα καινούριο στάδιο. Από τις 15 Ιουλίου και μετά η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και μάλιστα ίσως μοναδική στην ιστορία. Διότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε εναντίον του, των πραξικοπηματιών. Ο Μανώλης ε, γνωρίζει την, τι σημαίνει πραξικόπημα και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς επηρεάζει ένα πραξικόπημα μια χώρα. Όμως να σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου το έζησα και εγώ ο ίδιος προσωπικά. Γύρω στις 10 το βράδυ ε, άρχισαν να πετάνε αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι μας ε, κατάλαβα ότι κάτι κακό συμβαίνει. Άνοιξα την γερμανική τηλεόραση και είδα ειδήσει. Αναφερόταν ότι ε, στρατιωτικά γήματα έκλεισαν την κυκλοφορία στις γέφυρες της ε, Κωνσταντινούπολης πάνω από το Βόσπορο. Κατάλαβα ότι γίνεται πραξικόπημα. Πήρα τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου και ε, βγήκα στην κεντρική πλατεία της Άγκυρας. στο δρόμο μου τηλεφώνησε ένας συνάδελφος και με κάλεσε στην ε, Εθνοσυνέλευση, στη Βουλή μας. Εκεί μου είπαν αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να στείλουμε μηνύματα προς την κοινή γνώμη. Εκείνη την ώρα ήδη γίνονταν συγκρούσεις στους δρόμους. Εγώ άλλαξα δρόμο, πήγα στο κοινοβούλιο μαζί με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γύρω στα μεσάνυχτα ανοίξαμε το κοινοβούλιο και δηλώσαμε ότι ζούμε ένα πραξικόπημα που προσπαθεί να διασαλεύσει τη συνταγματική τάξη. Το είπαμε, το δηλώσαμε και, είπαμε ότι κινδυνεύει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία μας. Ξεκίνησαν όμως εκείνη τη στιγμή επιθέσεις από αέρος. Και κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών δεχτήκαμε τρεις φορές πλήγματα στο Κοινοβουλίο οι επιθέσει από αέρο αυξανόντουσαν. Οπότε ε, καταφύγαμε στο Κρυσφύγετο και συνεχίσαμε να δουλεύουμε εκεί. Δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαι βουλευτής, δεν είχα δει ποτέ επιθέσεις στο Κοινοβούλιο. Ε, επίθεση έγινε και εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου. και από αεροπλάνα και από ε, ελικόπτερα. 241 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, ή τη σωματική τους ακεραιότητα από αυτές τις επιθέσεις. αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της κατάστασης. Είδαμε πτώματα, είδαμε διαμελισμένα κορνιά και 2.000 άτομα τραυματίστηκαν, καταστράφηκαν πολλά κτίρια, ε, βομβαρδίστηκε το Προεδρικό Μέγαρο και η Βουλή όπως σας είπα. Σε ένα μόνο κτίριο έχασαν τη ζωή τους 50 άτομα. Δεν είναι ένα απλό στρατιωτικό πραξικόπημα, είναι ένα πραξικόπημα από μια συγκεκριμένη οργάνωση των γκουλενιστών συγκεκριμένα, ε, μέσα από το σύστημα, μέσα από το κράτος. Εδώ και 40 χρόνια ε, οι γκυλενιστές ε, έχουν ενταχθεί στον κρατικό μηχανισμό και στις ε, τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Και αυτοί διοργάνωσαν το πραξικόπημα. Η τρομοκρατική αυτή οργάνωση πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι. Εδώ και 40 χρόνια και δημοσίως αλλά και σιωπηρά ε, ε, έχουν ε, μπει στις, στο κράτος, στο δικαστικό σώμα, στην αστυνομία, στο στρατό, στην εκπαίδευση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην εκπαίδευση ιδιαίτερα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, με δημόσιο και διαφανή τρόπο, τρόπο χωρίς να το κρύβουν σε άλλες δημόσιες ε, υπηρεσίες με κρυφό τρόπο. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν μέσα στο κράτος μια παρακρατική οργάνωση ε, και με παράνομο τρόπο προωθούν τους δικούς τους ανθρώπους σε διαγωνισμούς ε, στρατιωτικών ακαδημιών ή αστυνομικών ακαδημιών. Ε, επίσης ε, χρησιμοποιούν τον εκβιασμό. Ε, πολλές ε, φορές δημιουργούν ψεύτικα πιστήρια αποδεικτικά στοιχεία για να εκβιάσουν συγκεκριμένους πολιτικούς. Κασέτες, βιντεοκασέτες και τέτοια. Οπότε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου δεν είναι ένα σύνθεση πραξικόπημα. Δεν είναι ένα από αυτά που είχαμε δει στο παρελθόν. Είναι μια τρομοκρατική δράση, μια δράση τρομοκρατικής οργάνωσης. Μετά τις 15 Ιουλίου ε, με τη διασάλευση της τάξης το χρειάστηκε να πολεμήσουμε αυτά τα στοιχεία. Ο πρόεδρος μας χρησιμοποίησε το άρθρο 120 ε, του συντάγματος και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, αυτή η κατάσταση προβλέπεται από διεθνείς συμφωνίες, όχι μόνο από το δικό μας σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο άρθρο 15 προβλέπει αυτή την κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Μου δίνετε πέντε λεπτά. Δύο. Είναι πολύ δύσκολο να σας διηγηθώ όσα έχουν συμβεί στην Τουρκία σε 5-6 λεπτά. Θα προσπαθήσω πάντως. Το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης ε, ε, που βρίσκεται στην κυβέρνηση ε, δεν αρέσκεται στην κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ε, εμείς έχουμε κήρυξη σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην νοτιοανατολική Τουρκία, για παράδειγμα. Ε, για την ακρίβεια εμείς ήραμε καταστάσεις έκθεσης ανάγκης που υφίσταντο το 2002 όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση. Ε, καταστάσεις έκτακτης ε, ανάγκης έχουν κηρυχθεί και σε άλλες χώρες και στη Γαλλία για παράδειγμα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εμείς έχουμε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα μπορώ να σας πω. Παρ' όλα αυτά, δεν κηρύττουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εύκολα. Ακόμα και στην, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, μετά από τέσσερις ώρες είχαμε άρει όλα τα μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ε, τέτοια κυβέρνηση, τέτοια χώρα είμαστε. Ε, ίσως αν μου κάνετε ερωτήσεις να σας δώσω απαντήσεις, αλλά στην εφαρμογή της κατάστασης έκθεσης ανάγκης θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Πρώτον, ε, βασιζόμαστε στις διατάξεις του συντάγματος. Στα άρθρα 120 ε, και 15 του συντάγματος. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ε, Επίσης βασιζόμαστε στο άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεύτερον, η, εθνική μας, η Εθνοσυνέλευσή μας ψηφίζει, ψήφισε και ψηφίζει όλες τις αποφάσεις για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει δικαίωμα να απορρίψει ή να τροποποιήσει μια τέτοια απόφαση και η απόφαση παράτασης για τρεις μήνες ελήφθη από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση πάλι. Μας υποστηρίζει η κοινή γνώμη. Ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαστε σε στενή συνεργασία μαζί τους. Ε, με πιέζει η κυρία ε, Πρόεδρος να τελειώσω. Υπάρχει το θέμα της ε, ελευθερίας έκφρασης. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο γιατί δεν έχω χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που χρειάστηκε να σας πείσω για το θέμα χρόνου, αλλά έχω πολλές ερωτήσεις και πρέπει θεωρητικά να τελειώσουμε σε 11 και είναι 11 παρά 1. Να πάμε 6 και τέταρτο τουλάχιστον. Έχω πολλές ερωτήσεις από συναδέλφους ομάδα αν συμφωνείτε και με τα υπόλοιποι. Αλλιώς θα μπορέσουμε να έχουμε την απάντηση του Υπουργού. Και έχουμε τη συζήτηση μετά αφού ολοκληρώσει ο Υπουργό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αναπολιτική ομάδα και μετά θα δούμε τι περιθώριο έχω για τους υπολοιπούς. Ο κ. Μπουσόη καταρχάς. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Uh, uh, Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Ρωτάει η πρόεδρος αν υπάρχει μετάφραση για τον Τούρκο Υπουργό. Τρεις ανησυχίες σχέση με την κατάσταση μετά από το πραξικόπημα και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πραξικόπημα το ίδιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε πληροφορίες ότι αυτοί που έχουν συλληφθεί από την κατ' Ιουλίου και μετά δεν μπορούν πλέον να έχουν υπεράσπιση. Δεν μπορούν να έχουν δικηγόρους, γιατί δικηγόροι επίσης έχουν συλληφθεί και αυτοί που δεν έχουν συλληφθεί ε, ε, ζουν υπό εκφοβισμό. Δεύτερο, εκτός από τις μικρές εταιρείε, πάνω από 300 ε, εταιρείε έχουν εθνικοποιηθεί είναι πάνω από 15 δισεκατομμύρια, εκα, ε, δισεκατομμύρια. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η κυβέρνηση της Τουρκίας και υπάρχουν επίσης και εκθέσεις από αξιόπιστα Ινστιτούτα όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Human Rights Watch ότι υπάρχει, υπάρχουν ε, εκτεταμένα περιστατικά βασανιστή, βασανιστήριων στους ε, κρατούμενους, κάποιοι από τους οποίους έχουν πεθάνει μέσα στις φυλακές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Παντσέρη. Μια παρατήρηση σύντομη και μια ερώτηση. Εσείς εφαρμόζετε το άρθρο 15 της σύμβασης. Όμως το άρθρο 15 της σύμβασης προβλέπει ότι δεν θα πρέπει επουδενή να παραβλέπονται τα άρθρα 2, 3, 4 και 7 της ίδιας της σύμβασης. Και επειδή ακριβώς υπήρξαν καταγγελίες σοβαρές για βασανισμούς και δολοφονίες έχετε πρόβλημα και θα πρέπει να δώσετε απάντηση στη διεθνή κοινότητα εκτός από αυτή την υποεπιτροπή. Yes, uh, Mr. Dank u, uh, meneer de uh, onderminister. Ευχαριστώ. Υφυπουργέ, κοίταξε τα νούμερα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, διαβάζω ότι υπάρχουν 6.000 συλλήψεις, πολύ κρατικοί υπάλληλοι, 8.000 αποφυλακίσεις αστυνομικών και 7.000 δικαστές ανακρίθηκαν πολλοί ε, κρατούμενοι δεν έχουν πρόσβαση σε νομική παράσταση. Υπάρχουν εκθέσεις ε, για βασανιστήρια και η αντίδραση των ε, εθνικών αρχών μου δεν μου φαίνεται ανάλογη προς το πρόβλημα. Υπάρχει καταπίεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρκετές εφημερίδες έχουν κλείσει και κανάλια. Πολλοί δημοσιογράφοι συλλήφθηκαν και η απειλή αυτή σκιάζει όλη τη χώρα. Στη χώρα μου στο Βέλγιο υπάρχει μια εφημερίδα η Ζάμαν Φαντάχ, η βελγική έκδοση της Ζάμαν και αυτή παρουσιάζει πλέον ε, τους γιουλενιστές ως τρομοκράτες παράνομη βία, γίνεται χρήση παράνομης βίας που αποσκοπεί ε, στο να θυματοποιήσει τους πολίτες. Αυτό το ε, επιχείρημα που χρησιμοποιείτε, μήπως είναι μια πρόφαση για να ασκήσετε αυτά τα... Ευχαριστώ κύριε Ο κύριος συγγνώμη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά το πραξικόπημα, την αποτυχημένη απόπειρα. Πολλές, πολλά πολιτικά κόμματα, όπως και το δικό μου, καταδικάσαμε αυτή την παράνομη δράση ή πράξη και σωστά το κάναμε. Υπάρχουν όμως διάφορες συλλήψεις διαφόρων αξιωματούχων, καθηγητές, πανεπιστημιακοί κτλ. Δεν είναι μόνο περιστατικά αυτά, χιλιάδες. Πώς εξηγείται λοιπόν το γεγονός ότι καθηγητές και δάσκαλοι είχαν εμπλακεί στο πραξικόπημα σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα κατά του κράτους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ποια αρχή αναλογικότητας εφαρμόστηκε αφού λήφθηκε αυτή η απόφαση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ε, κυρία Πρόεδρε, απλώς για να κάνουμε την συνεδρία πιο σύντομη, οι ερωτήσεις μου έχουν υποβληθεί και νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσω εδώ. Ευχαριστώ. Sí, eh, señor Ευχαριστώ, κύριος Χάμς. Ja, ich möchte als Señora Harms, Ja, ich möchte als erstes noch θα ήθελα να τονίσω ότι όταν μιλάω με συνέλευση από το τουρκικό κοινοβούλιο και εκπροσώπους του ΑΚΠ κρίνουν ε, φυσικά ότι καταδικάζουν το πραξικόπημα, αλλά ότι ανησυχούν ταυτόχρονα για αυτά που έχουν γίνει και για το αν η Τουρκία μετά από το πραξικόπημα θα είναι να έχει κράτος δικαίου, να παρέχει κράτος δικαίου. Αυτό που είπε ο κύριος Ντεμές Μέκερ ε, το επισημαίνω και εγώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ανησυχίες αν μπορεί να εγγυηθεί η Τουρκία το κράτος δικαίου και ένα πρόβλημα μεμονωμένο που θέλω να τονίσω για τους συλληφθέντες και τους κρατούμενους. Ανάμεσα τους υπάρχουν πολλοί δικηγόροι, πολλοί δικαστές που δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα σε νομική παράσταση, σε ατομική δίκη η οργάνωση ανεξάρτητων δικαστών απαγορεύτηκε στην Τουρκία και θέλω να μάθω από εσάς εδώ σήμερα πώς οι δικαστές στην Τουρκία στις δίκες που προετοιμάζουν θα μπορέσουν να σκίσουν ανεξάρτητα το έργο τους όταν αντιμετωπίζουν την απειλή να βρεθούν εν μία ανοιχτή στη φυλακή επειδή προσπάθησαν να λάβουν μια ανεξάρτητη απόφαση. και ε, απειλούνται με την κατηγορία της τρομοκρατίας αυτή δικαστής. Πώς μπορούν να αποφασίσουν ανεξάρτητα σε μια τέτοια κατάσταση όπου τους ασκείται δίωξη, ασκείται δίωξη γενικότερα στην, στον κλάδο της δικαιοσύνης. Voy a Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο εκπρόσωπο πολιτικής ομάδας. Λυπάμαι, αλλά δεν θα δεχτώ άλλες ερωτήσεις. Θα απαντήσω ο Υφυπουργό. Ήδη έχουμε περάσει τον χρόνο το διαθέσιμο κατά πολύ και έχουμε στη συνέχεια τη συζήτηση όπου μπορείτε να λάβετε το λόγο όλοι. Αν όμως δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους, δεν θα απαντήσει ο Υφυπουργό. Ο κ. Παπαδάκης τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βασικά θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα σε σχέση με τη στάση της ε, κυβέρνησης της Τουρκίας και το ζήτημα της αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης. Το να φτάνει ε, μια κυβέρνηση να αμφισβητεί διεθνώς αναγνωρισμένες και συμφωνημένες ε, συνθήκες, όπως η συνθήκη της Λοζάνης, που προϋποθέτει αμφισβήτηση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη πράξη, ε, την οποία θέλουμε να καταδικάσουμε και βέβαια πρέπει να διαμηνήσουμε ότι αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη. Ακριβώς γιατί σε μια ιδιαίτερα έφλεκτη ε, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στη Συρία, την οποία εκτός από τις επιθέσεις των ε, υπεριαλιστών της, ε, των ΗΠΑ και, της, ε, και όλων των άλλων κρατών που εμπλέκονται στην όλη αναμέτρηση και η Τουρκία ε, ήδη έχει εισβάλει και στο Ιράκ. Το λέμε αυτό λοιπόν σε τέτοια επικίνδυνη περίοδο η ε, ανακοίνηση τέτοιων ζητημάτων, τέτοιων ανύπακτων ζητημάτων, συμφωνημένων ζητημάτων ε, στην ευρύτερη περιοχή είναι σε βάρος των λαών και ανακοινεί και εθνικιστικά μίση και βέβαια από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να τοποθετηθείτε υπεύθυνα και συγκεκριμένα. Και βέβαια παίζει ε, ρόλο και ιδιαίτερη ευθύνη έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που με τη στάση τους επί της ουσίας, ε, τη στάση των ίσων αποστάσεων όλο αυτό το διάστημα δημιουργούν έδαφος για τέτοια επιθετικότητα και προκλητικότητα. as your, as your best, ε, Κύριε Υπουργέ, βάλτε τα νατά σας, ό,τι μπορείτε. Παρακαλώ. Ε, τη νύχτα της 15ης ε, Ιουλίου, ε, τι, ποια ήταν τα αισθήματά μου, αναρωτιέμαι πολύ συχνά. Δεν φοβήθηκα. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα. Αυτό που αισθανόμουν ήταν ντροπή. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Τουρκία είναι μια ανεπτυγμένη χώρα και στην οικονομία και στη δημοκρατία. Μπορεί να έχει αδυναμίες η δημοκρατία, μπορεί να έχουμε προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα 15 τελευταία χρόνια διανύσαμε πολύ μεγάλη απόσταση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το πούν όλοι, να το δεχτούν. Δεύτερον, δεύτερος λόγος ντροπή. Δεν άκουσα τίποτα από εδώ από την Ευρώπη, καμία αντίδραση. Ε, δεν τοποθετηθήκατε υπέρ του κράτους δικαίου αμέσως. Δεν τοποθετηθήκατε υπέρ της Τουρκίας αμέσως. Περιμέναμε δύο-τρεις μέρες, δύο-τρεις εβδομάδες για να ακούσουμε αντίδραση υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό με έκανε να νιώσω ντροπή. Στο να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τι συλλήψει των ε, δικηγόρων και της, ε, του μη διορισμού δικηγόρου. Όλοι έχουν δικαίωμα σε υπεράσπιση. Όλοι όσοι έχουν συλληφθεί έχουν προσαχθεί σε δικαστή και έχουν δικηγόρο. Ε, με μια απόφαση περασμένη εβδομάδα ε, ε, δημιουργήσαμε μια επιτροπή παραπώνων ε, που συμμετέχουν όλοι οι αναπληρωτές υπουργείων, όλων των υπουργείων ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να εξετάσουμε οποιοδήποτε ισχυρισμούς αδικίας ή μεροληψίας. Δεν είναι εύκολο να καταλάβετε το πραξικόπημα αυτό. Δεν ζήσατε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Δεν είδατε τη βουλή σας να βομβαρδίζετε. Είναι δύσκολο να τα βάλετε αυτά με το μυαλό σας. Άλλωστε δεν έχετε και τέτοια παράδοση. Θα ήθελα όμως Ε, θα ήθελα να ρωτηθείτε όμως, με αυτές τις ε, διαμαρτυρίες σας ε, υπερασπίζεστε τα δικαιώματα και τη μνήμη των 241 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους. Υπερασπίζεστε το δίκιο τους. Στο όνομα του κράτους δικαίου δεν βλέπετε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει στην Τουρκία. Υπάρχουν άνθρωποι πράγματι που τέθησαν σε αργία και συνελήφθησαν. Όμως, ο δικαστικός μηχανισμός λειτουργεί. Ε, δεν αφαιρέσαμε το δικαίωμα σε πρόσβαση σε δικηγόρο από κανέναν. Επίσης, ε, είμαστε ανοιχτοί σε διεθνείς παρατηρητές. Και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις βασανιστήριων. Ε, εμείς δώσαμε τέλος στα βασανιστήρια από όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2002. Ε, και γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία 15 χρόνια, ε, έχει βγει από την ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Δεν δεχόμαστε καν καταγγελίες γι' αυτό δεν υπάρχουν καταγγελίες. Τώρα, για οποιαδήποτε η καταγγελία για αυτή την εποχή θα, την θα τη διαρευνήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Παντζέρη και το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλοι όσοι έχουν υπογράψει τη σύμβαση μπορούν να το επικαλεστούν και δίνει το δικαίωμα να ανασταλούν συγκεκριμένα άρθρα. Και στην ε, Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες ε, μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις έγινε τέτοιου είδους αναστολή, χρησιμοποιήθηκε αυτό το άρθρο προκειμένου να προστατευθούν οι χώρες αυτές από διασάλευση της τάξης. Όπως σας είπα, η δράση μας βασίζεται και στο Σύνταγμα, άρθρα 120 και 15, και στο άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, η κοινή γνώμη μας υποστηρίζει, η αντιπολίτευση μας στηρίζει σε αυτή τη χρήση του άρθρου. Σε οκτώ χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μετρήσαμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το άρθρο. Σε Ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, να σας πω το εξής. Ίσως για να καταλάβετε καλύτερα να σας πω το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίστηκαν το πραξικόπημα στην Τουρκία, ο, ο, ο, επικεφαλής τους ήταν ε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σακάρια. Του Σακάριου δηλαδή. Ε, ε, ε, Ήταν τέτοια η οργάνωση του πραξικοπήματος που κάθε ομάδα που συμμετείχε δεν ήξερε τι υπήρχε από πάνω της. Ε, Ήταν μια πυραμιδωτή οργάνωση. Εκείνο το βράδυ Στα τάγκς, μέσα στα τάγκς ε, υπήρχαν άνθρωποι της οργάνωσης των κυλενιστών και πριν μερικές μέρες πριν το πραξικόπημα ε, ε, κάποιος ε, από τους γκουλενιστές ε, που ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει θα ήθελα να είμαι συνταγματάρχης για να βοηθήσω καλύτερα τη χώρα μου. Καταλαβαίνετε που αποσκοπούσε. Πολλά μέσα μαζική ενημέρωση, πολλοί δημοσιογράφοι στήριξαν αυτή την οργάνωση των Κιλίνστον και θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην κοινωνία. Η διαδικασία, όμως η δικαστική διαδικασία θα γίνει κανονικά. Ε, οι κανόνες τηρούνται και θα τηρηθούν και όποιοι δεν είναι υπεύθυνοι δεν θα καταδικαστούν και θα απελευθερωθούν. Οι δε ένοχοι θα τιμωρηθούν όπως πρέπει. Για την Λοζάνη για τη συνθήκη της Λοζάνης. Ε, ε στην ε, Τουρκία αυτό που συζητείτε αν είναι αν η συνθήκη της Λοζάνης ήταν επιτυχία ή αποτυχία για την Τουρκία. Ε, αυτό είναι εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία, δεν έχει σχέση με την εξωτερική μας πολιτική. Ε, η συμφωνία ισχύει. Ευχαριστώ. Ωραία. Λέει πρόεδρο, δεν είναι η τελευταία συζήτηση, ούτε η τελευταία συνεδρίαση για την Τουρκία. Η παρουσία του Υφυπουργού ήταν ξαφνική. Τώρα έχουμε μία ακρόαση με εμπειρογνώμονες και με άτομα που προασπίζονται την ελευθερία του κράτους δικαίου στην Τουρκία και σα καλώ να παραμείνετε στην αίθουσα γιατί ήρθαν οι προσκεκλημένοι μα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υφυπουργέ. Vamos a proseguir, por favor. Ahora está con... Θα συνεχίσουμε. Ήρθε και ο κύριος Μπροκ τώρα. Θα προσπαθήσουμε να πάμε γρήγορα για να μπορέσετε να μιλήσετε όλοι, γιατί πολλοί βεβαίως δεν έλαβαν το λόγο προηγουμένως. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχουμε σήμερα αυτή την ακρόαση. Όπως γνωρίζετε, με την Κέτη Πέρι, μετά από το πρακτικό που πήγαμε στην ε, Τουρκία, με την Κάθη Πέρι, και εκφραστήκαμε ενάντια στο πραξικόπημα και αυτό ήταν το σωστό. Αυτό το πραξικόπημα μια στρατιωτική παρέμβαση σε ένα δημοκρατικό κράτος που απείλησε με βομβαρδισμό το κοινοβούλιο και που παρατρίχα 150 βουλευτές θα σκοτώνονταν αν επιτύχανε αυτή η απόπειρα βομβαρδισμού. Η κριτική που στην εσωτερική ε, πολιτική για την ελευθερία της έκφρασης ε, είναι ένα θέμα, όμως προτιμούμε να συζητάμε με μια δημοκρατική κυβέρνηση παρά με μια στρατιωτική κυβέρνηση, μια δικτακτορική κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα του πραξικοπήματος ε, μάλλον το πραξικόπημα ήταν αποτέλεσμα υπόγειων δομών που υπήρχαν και τις οποίες δεν γνώριζε και είχε υποτιμήσει η τουρκική κυβέρνηση. και που ε, διαμορφώθηκε μακροπρόθεσμα και που από κοινού με, την, ε, ε, με το κίνημα του Γκιουλέν απειλούσε να οδηγήσει αστάθεια την Τουρκία. Αυτές οι παράλληλες δομές, όπως είπα και πριν, και με τις οποίες παράλληλες δομές η τουρκική κυβέρνηση για πολύ καιρό συνεργάστηκε για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν αποτελεί όμως αυτό δικαιολογία για το πραξικόπημα. Υπήρξε αυτή η συνεργασία για να εκτοπιστούν οι κεμαλιστές ουσιαστικά. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και ένα τρίτο σημείο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια Τουρκία που είναι με το μέρος της Δύσης και να μην κατευθυνθεί σε λάθος πορεία, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Αυτό που συμφέρει τους Τούρκους μας συμφέρει και μας όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά και ως στρατηγική παγκόσμια. Αυτό μας σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τα πάντα. Κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά θα πρέπει να τηρηθούν όπως και από τις άλλες χώρες γιατί θα πρέπει να πετύχει τα στάνταρ, τα πρότυπα ενώ μια υποψήφια χώρα η Τουρκία αν θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει αυτά τα πρότυπα της ελευθερίας του λόγου, του κράτους δικαίου κτλ. Και έχω την αίσθηση ότι τους τελευταίους μήνες οπισθοδρομήσατε σε σχέση με όλα αυτά. και μέχρι που σκεφτεί να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 24. Αυτό όμω είναι μια άλλη συζήτηση, υπό τα οποία θα υπήρχε και μια πολύ πιο στενή, ένα πολύ πιο στενό screening. Πρέπει να αντιρευνήσουμε το θέμα του κράτους δικαίου, να δούμε το στάτους της Τουρκίας ως προς την ικανότητα προσχώρησης. και να κάνουμε μια αποτίμηση του πραξικοπημάτος. Βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλές απολύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, συλλήψεις και την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Γιάνγκλαντ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κύριος Γιάνγκλαντ που ήταν στην, Ευρώ, ε, στην Τουρκία και που έκανε προτάσεις και που έθεσε το θέμα του κράτους δικαίου σε σχέση με το θέμα της ε, αναλογικότητας. το δικαίωμα σε νομική παράσταση που πρέπει να έχουν οι κρατούμενοι και όλα αυτά επίσης μας απασχολούν και θεωρώ ότι είναι ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Συμβούλιο, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να μπορέσει να αποδείξει και να πετύχει αυτό το πρότυπο, είναι υποχρέωση και θα ήταν σωστό να διερευνήσουμε την ποιότητα και την δυνατότητα που έχει η Τουρκία για την προσχώρηση και να εξασφαλίσουμε και την ύπαρξη κράτους δικαίου με ενδιαφέρει πολύ να μάθω την άποψη των εμπειρογνωμόνων. Πού υπάρχουν ελλείψεις, πού υπάρχει πρόοδος και τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενους μήνες, όπου θα υπάρχουν ε, συζητήσεις και διάλογος με τους ε, Τούρκους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Μπροκ. Ίσως ο κύριος Κεφαλογιάννης να θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Βαλενθιάνου και τον κύριο Μπροκ που είναι εδώ σήμερα για αυτή τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Η συνεργασία μεταξύ και ουλευτικών επιτροπών και υποεπιτροπών είναι πολύ σημαντική επειδή χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο συνδυαστικά εμπειρία και πόρους. Συνεδριάζουμε τρεις φορές ετησίως με βουλευτές από την Τουρκία. Μετά από αυτά που έγιναν όμως πρόσφατα αναβάλαμε τις συνεδριάσεις μας για τη συνέχεια αλλά με τον κύριο Σαχίν και τον πρόεδρο μας τον κύριο Κονκάρ ολοκληρώσαμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίασή μας που θα γίνει στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επομένου. Είναι σημαντική συζήτηση λοιπόν σήμερα για το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Ελπίζω να την συνεχίσουμε στην Άγκυρα και ζητήσαμε την άδεια από το Κοινοβούλιο να διεξαχθεί συνάντηση αυτή στην Τουρκία ακριβώ για να υπογραμμίσουμε την σημασία της Ευρώπης στην σταθεροποίηση της Τουρκίας. Γιατί ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που θα ήταν καλό να είχαμε αυτή τη σταθερότητα. Και μιας και εμείς και ο Υπουργό εδώ για την συνθήκη της ε, λοζάνη πολυμερή συμφωνία που υπογράφηκε από διάφορε χώρες. Τουρκία, Ελλάδα, αλλά Βουλγαρία, αλλά Γερμανία, ΙΠΑ, Ιαπωνία και άλλες χώρες που αποτελεί τον πυρήνα της ύπαρξης του νέου τουρκικού κράτους ως εξέλιξη του Οθωμανικού τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό για σταθεροποίησε την περιοχή μετά από τα αρχές δεκαετιών. Καθόρισε τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως επίσης και της ε, Τουρκίας με την ε, Συρία και άλλες χώρες. Και, και κυρίως βεβαίως ρύθμισε το θέμα του Ελισπόντου, το οποίο ρύθμισε την κίνηση την εμπορική για πολλά χρόνια. Οπότε πρέπει να κάνουμε συζητήσεις περαιτέρω για το κεκτημένο και για το πώς η Τουρκία θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δυστυχώς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα χρόνου, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ την κατανόησή σας. Σας παρακαλώ να είστε περιεκτικοί, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Βουλή είμαστε, πρέπει να μιλήσουν οι βουλευτές και οι βουλευτίνες. Καταρχάς, σύντομα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αμπέρ Ντεβιολέ, γιατί όπως είπε ε, ο κύριος Μπροκ, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ένα σημαντικό ρόλο και από εκεί προέρχεται ο κύριος Ντεβιολέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που καλέσατε το Συμβούλιο της Ευρώπης να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση σήμερα. Ο κ. Σαββασόγλου θα μιλήσει και στην ε, συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο και ο Γενικός Γραμματέας επειδή χρειάστηκε να πάει εκεί, μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω εδώ στην ε, ακρόασή σα και να σα ενημερώσω για την συνεργασία που έχουμε με την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Ο διάλογος με την Τουρκία για αυτά τα θέματα βασίζεται σε τρεις κύριες πρωτοβουλίες. πρωτοβουλίες. Καταρχάς έχουμε μια ομάδα εργασία για την χάρτα της Ένωσης και την εφαρμογή της. Νομοσχέδια που αφορούν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μετά εποπτεία θεμάτων που αφορούν βεβαίως βασανιστήρια, φυλακής κλπ. Καταρχάς, για την απόφαση των δικαστηρίων για την Τουρκία. Έχουμε μια άτυπη ομάδα εργασία, η οποία συγκροτήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του 2015 σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνη τη Τουρκία. Η τελευταία συνάντηση έγινε τον Ιούνιο φέτο και επικεντρώθηκε σε περιορισμού όσον αφορά την ελευθερία έκφραση, το άρθρο 10 του, της, ε, της Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 11 επίση, ε, ελευθερία συναθρίζεστε, και αυτές οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ε, ερμηνεία της νομοθεσίας σε σχέση με την τρομοκρατία, τρομοκρατικές ε, πράξεις, ποινικό κώδικας, οικονομικός κώδικας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έγινε και σύμφωνα με αυτό που λένε και τα διεθνή δικαστήρια για παραβίασης παραβίασεις των άρθρων 10 και 11 και τις αποφάσεις ε, απόφαση που αφορούν αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά εξετάζονται από τις, από τις τουρκικές αρχές. Στις συζητήσεις μας πάντως θέλουμε να επικεντρωθούμε βεβαίω τις εκτελέσεις των αποφάσεων των δικαστηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποτρέψουμε βεβαίω την περαιτέρω παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δεύτερον, συνεργασία για τα νομοσχέδια που αφορούν την κατάσταση, την εκτακτή κατάσταση μετά το πραξικόπημα. Δεχτήκαμε ένα αίτημα για παρέκκληση από την Τουρκία είπε το άρθρο 15.3 της ε, χάρτας. Αυτή η εξαίρεση έλαβε χώρα αμέσως και κοινοποιήθηκε βεβαίως όλα τα υπογράφοντα μέλη της ε, σύμβασης. Όπως λέει το άρθρο 15, οι τουρκικέ αρχέ μετά ενημέρωσαν την, τον Γενικό Γραμματέα για τα μέτρα που λήθησαν υπό το καθεστώς έκτακτης ε, ανάγκης. Εργαζόμασταν λοιπόν σε, με, σε, με τρεις διαφορετικούς τρόπους στα νομοσχέδια που έθέσε η Τουρκία. Καταρχάς τα λαμβάνουμε, ξεκινάμε ένα διάλογο και αυτό οδήγησε σε μια συνάντηση που είχαμε στις 2 του Σεπτέμβρη συνάντηση με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας. Είχαμε μια δεύτερη συνάντηση στην Άγκυρα και αυτή το Σεπτέμβριο. Συνεχίζονται οι διαβολεύσεις με στόχο να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται υπό το νομοσχέδιο θα πρέπει να σέβονται το κριτήριο αναλογικότητας και θα πρέπει βεβαίως να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κυρίως ε, η συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλη μία πρωτοβουλία ε, αφορά την Επιτροπή Βένης που προσκλήθηκε ε, στην, στην Εθνοσυνέλευση για να δει αυτά τα νομοσχέδια υπό το φως των αποφάσεων που λέγαμε προηγουμένως. Θα υιοθετηθεί ε, η γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής από το Συμβούλιο της Ευρώπης το Δεκέμβρη. Επίσης, έχουμε και το θέμα της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας στην Τουρκία. Η Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει αυτή τη βδομάδα στη Βενετία για αυτό το ζήτημα, για την άρση της ε, κοινοβουλευτικής ασυλίας. Για τα νομοσχέδια, η Επιτροπή μας ή μάλλον επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κ. Μουστινής, τον Οκτώβρη δημοσίευσε ένα έγγραφο που αφορά την επισκεψή του στην Τουρκία και παρουσιάζει τις απόψεις του Επιτρόπου που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχέση με την κατάστασή τους. Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στην Τουρκία, η Επιτροπή για την, ε, για την Αποτροπή Βασανιστήριων επισκέφθηκε την Τουρκία 29 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτέμβριου ώστε να εξεταστεί εξεταστούν συνθήκες κράτησης και μεταχείριση των κρατουμένων σε σχέση με το πρόσφατο πραξικόπημα. Η αντιπροσωπεία είχε ιδιωτικές επαφές στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Ε, τελειώνεται λέει πρόεδρος στείλαμε την ε, έκθεση την οποία θα δημοσιεύσουμε, θα δημοσιεύσουμε τη στείλαμε και στις τουρκικές αρχές για διαβούλευση και να τελειώσω για τα υπόλοιπα θέματα, με τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου και να πω ότι είχαμε σημαντική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεβέντ Κορκούτ έχει το λόγο τώρα, είναι καθηγητής, ειδικό ε, συνταγματικού δικαίου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. going to speak in... Θα μιλήσω στα τουρκικά. Αν όμως ε, χρειάζεστε διευκρινήσεις, επεξηγήσεις, μπορώ να χρησιμοποιήσω και την αγγλική αργότερα. Ε, ε, θα μιλήσουμε για την κατάσταση μετά το πραξικόπημα. Την απόπειρα πραξικόπηματος, να το πούμε καλύτερα. Ε, αλλά ε, πρέπει να δούμε και την ανθρώπινη διάσταση. 241 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Από πλευράς ε, κράτους δικαίου, ε, θα πρέπει να γίνει όλη η προσπάθεια προκειμένου να διαλευκανθούν τα γεγονότα και το πώς έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι και βέβαια πώς τραυματίστηκαν οι τραυματίες. Ε, υπάρχουν ευθύνες οι οποίες θα πρέπει να καταδειχθούν από το δικαστικό μας σύστημα. πώς οργανώθηκε η απόπειρα πραξιοποίηματος, ποιοι ήταν υπεύθυνοι. Όλα αυτά θα πρέπει να διαλευκανθούν. Ένα κράτος δικαίου έχει, οφείλει να το κάνει αυτό. Το αναμένουν οι πολίτες μας και θα πρέπει να το πράξουμε. Ή τώρα, είναι απολύτω απαραίτητο γι' αυτό να ενημερώνει το λαός. Πλήρης ενημέρωση. Απ' την άλλη μεριά, ένα κράτο δικαίου, κάνοντας αυτή τη διαλεύκανση, θα πρέπει να προσέχει ορισμένα πράγματα. Και γι' αυτό το ζήτημα ε, γίνεται πολλή συζήτηση. Και όπως είπε ο εκπρόσωπος της Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, προετοιμάζεται και μια έκθεση για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να δούμε το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα τη διαδικασία. Ε, το πλαίσιο της έκθεσης, για το πλαίσιο της έκθεσης θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Το, ε, Όπως γνωρίζουμε, πάρα πολλοί κρατικοί υπάλληλοι τέθησαν σε αργία ή απολύθησαν τα τους τελευταίους δύο-δυόμιση μήνες. Αυτό το γεγονός δεν είναι κάτι καινούριο την Ευρώπη. Ε, υπάρχουν αποφάσεις τέτοιου τύπου στο παρελθόν. Σε περίπτωση μετάβαση. δημοκρατικής ε, ε, πολλές χώρες έχουν λάβει τέτοιου αποφάσεις σε θέση αργία δημόσιων λειτουργών. Στην Μακεδονία, για παράδειγμα, λέει ο Μιλτής, την Πολωνία κλπ. Όμως υπάρχουν νομικά θέματα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκφέρει άποψη. Και θα πρέπει να υπονομήσουμε το εξή. Ε, αυτά του τα μέτρα συνήθως ονομάζονται μέτρα εκαθάρισης. Και βασίζονται κανονικά σε τέσσερις αρχές. Οι κρατικοί πάλι που απολύονται θα πρέπει να απολύονται με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τον κάθε έναν από αυτούς και θα πρέπει να αποδειχθούν οι υπόνοιες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Τουρκίας θα πρέπει να αποδειχθεί ότι κάθε ένας από αυτούς ήταν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι εργαζόταν για τα συμφέροντά της. Δεύτερο, δεύτερη αρχή, δεύτερος όρος, θα πρέπει να τους, δοθεί πλήρη, να τους δίδονται πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης. Δυστυχώς, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση. Ε, δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην υπεράσπιση, αλλά και το ε, τεκμήριο αθότητας, το οποίο πλήττεται. Και ο τύπο στα μέσα ενημέρωση, αλλά και διάφορες δημόσιες ε, δηλώσεις ε, ε, τίνουν να υποδεικνύουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ήδη ένοχοι αυτοί που συλλαμβάνονται. Και αν απελευθερωθούν θα έχουν στιγματιστεί. Αν αθωωθούν δηλαδή θα έχουν στιγματιστεί. Δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να τηρούμε το, κριτήριο της, το τεκμήριο της αθότητας. Άλλος όρος. Θα πρέπει να ε, προασπιστούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Πολλοί υπάλληλοι χάνουν τα δικαιώματα κοινωνική του ασφάλισης όταν απολύονται. Αυτό πρέπει να γίνεται ότι είναι ότι για κάθε υπάλληλο θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο ντοσιέ, ιδιαίτερο φάκελο και να μην απολύονται ή να τίθενται σε αργία μαζικά από, ε, με βάση κάποιε λίστες. το, θα πρέπει να παραμείνουμε στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου και να ε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και το εξή. Το άρθρο 15 του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 15 ε, δεν προβλέπει την αναστολή της ίδιας της ε, σύμβασης. Ας το υπογραμμίσουμε αυτό. Ε, όλες οι δράσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές. Δυσανάλογες δράσεις και μέτρα ε, θα κριθούν και από τα τουρκικά και από τα διεθνή δικαστήρια. Το άρθρο 15 λοιπόν της ε, σύμβασης δίνει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ε, δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης των μέτρων, αλλά με τρόπο αναλογικό, όχι δυσανάλογο. Η αναλογικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση και σε κάθε περίπτωση. Όμως έχουμε δει πολλά μέτρα τα οποία είναι δυσανάλογα. Τέλος, τέλος αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Το πρόβλημα της Τουρκίας ε, θα πρέπει να ιδωθεί στο σύνολό του. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Τουρκία τα τελευταία 15 περίπου χρόνια δείχνουν ότι η κοινή γνώμη έχει στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θα πρέπει να βλέπουμε την κάθε περίοδο αποκομμένη από τις υπόλοιπες. Ε, ε, η μεταρρύθμιση του στρατού ήταν πολύ σημαντική. Ε, ε, θα συζητηθούν θέματα ανθεώρησης συντάγματος τον επόμενο καιρό, τις επόμενες εβδομάδες. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δημοκρατία. Οι θρησκευτικέ ελευθερίες, ε, η λειτουργία των θρησκευτικών αδελφοτήτων και των διαφορών δογμάτων είναι θέματα που επίσης πρέπει να συζητηθούν. Όποια και είναι τα προβλήματα της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και όλα τα όργανα. Λυπάμαι, λυπάμαι κύριε καθηγητά, πρέπει να σας διακόψω, αλλά ε, έχουμε άλλους τρεις ανθρώπους. Να... Και εσείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε όριμα τα πράγματα, οι προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως όχημα υπέρ ή κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ να αντιμετωπίσετε με οριμότητα την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που σας πιέζω, αλλά μας λείπει χρόνος και ο χρόνος εδώ δεν είναι αιώνιος. Ο κύριος Ιπραχήν Καπολούκη που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μαρμάρα στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα παρέμβω στα γαλλικά, όπως είχε προβλεφθεί. Ε, έστειλα και ένα κείμενο, εννέα σελίδων, ε, για να διανεμηθεί. Σε δέκα λεπτά προφανώς δεν μπορώ να σας διαβάσω το κείμενό μου. Ε, θα πάρω κι εγώ δέκα λεπτά όπως και ο συναδελφός μου και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη Θα ξεκινήσω με μια ε, φράση ε, ε, του Ζαν Μάρκ, του συνάδελφού μας, που, είναι ειδικευμένος στην Τουρκία. Τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου ε, απέτυχε μια απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία ε, ευτυχώς για τη δημοκρατία. Ε, είχα προετοιμάσει την παρέμβασή μου σε τρία, τρεις άξονες. Πρώτον, ε, το φαινόμενο της αποσυνταγματοποίηση που παρατηρείται στην συνταγματική μας ιστορία και πριν ακόμα το πραξικόπημα. Δεύτερον, η απόπειρα πραξικοπήματος και ε, μια έκκληση για την προάσπιση του κεντρικού πυρούνα των δικαιωμάτων ε, στην Τουρκία, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τρίτον, ε, τα νομοθετικά διατάγματα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στην Τουρκία μετά το ε, πραξικόπημα και οι σχέσεις τους με το κράτος δικαίου. Ε, πριν το ε, πραξικόπημα λοιπόν η αποσυνταγματοποίηση της συνταγματικής μας τάξης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει το εξής. Ότι εδώ και δέκα περίπου χρόνια συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, μια έμεση ή ρητή συμμαχία ανάμεσα στο κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης και το, τους γκυλενιστές. Και δεύτερον, η απομάκρυση η αλλίωση των συνταγματικών, της εφαρμογής των συνταγματικών αρχών με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό σταδιακά. Δύο συνταγματικέ διατάξει θα θέσω υπόψη σα. Η πρώτη αφορά τι θρησκευτικέ αδελφότητε και η δεύτερη αφορά την απαγόρευση τη πολιτική εκμετάλλευση τη θρησκείας. Οι θρησκευτικέ αδελφότητε δεν έχουν συνταγματικό καθεστώ στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά τέτοιου είδου δραστηριότητε μπορούν να γίνονται στο πλαίσιο του άρθρου 24 του συντάγματος που αφορά την θρησκευτική και ελευθερία και την ελευθερία συνείδησης. Σύμφωνα με το οποίο οι προσευχές ε, και οι θρησκευτικές τελετουργίες είναι ελεύθερες υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν με, τις, ε, με το άρθρο 14 του Συντάγματος όπως το άρθρο 17 της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή είναι το άρθρο που απαγορεύει την κατάχρηση του δικαίου. Και δεύτερη διάταξη στην οποία αναφέρθηκα, άρθρο 24, κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την θρησκεία ε, για τη διασάλευση της οικονομικής, ε, πολιτικής, ε, ε κοινωνικής και συνταγματικής τάξης. Εδώ γίνεται λόγος λοιπόν για την σχέση ανάμεσα στις ε, θρησκευτικές και το κράτος. Οι θρησκευτικές αδελφότητες παρέβησαν το άρθρο 24 και από την άλλη μεριά το κράτος, η κυβέρνηση μάλλον, ε, ε, έκανε το ίδιο διότι έφερε την θρησκεία, της θρησκευτικές αδελφότητες μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συσσαγωγικά μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών και τις συνταγματικές αναθεωρήσεις και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι το 2010 έγινε μια σημαντική συνταγματική αναθεώρηση σε συνεργασία με τους γκυλενιστές. Ε, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είχαν παρουσιαστεί ως συνταγματική επανάσταση για την αναδιάρθρωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εισαγγελέων και Δικαστών και του ε, α, Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε αυτή τη διαδικασία ε, ε επλήγησαν ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εμείς ε, κατηγορηθήκαμε, δικαστήκαμε στο ανώτατο δικαστήριο διότι είχαμε κατηγορηθεί ως γιουλενιστές. Αυτή η διαδικασία είναι συνεχής. και ε, αποτελεί ε, αλλίωση του συντάγματος. Και μετά την, τις τελευταίες εκλογές ε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο καινούριος πρόεδρος, ο κ. Σερντοάν, είχε πει ότι στόχος του είναι, μάλλον η εκλογή του σηματοδοτεί την μετάβαση σε ένα προεδρικό καθεστώς, σε μια προεδρική δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος έγινε μια δήλωση ε, από την ε, πρωτοβουλία Πρώτα Δημοκρατία στις 20 Ιουλίου συγκεκριμένα, τέσσερις ε, μέρες μετά. Είναι, περιέχει 15 άρθρα και λέει καταδικάζουμε την απόπειρα πραξικοπήματος, καλούμε τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν το κράτος δικαίου. Αυτό είναι ο τίτλος της δήλωσης. Θα περιοριστώ στο να σας διαβάσω μόνο την αρχή παριθμό 13. Η ο πρώτος όρος για την επιτυχία του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Τουρκία είναι η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία να εξασφαλίσουν τη συνένεση σε ό,τι αφορά το σεβασμό του συντάγματος και τη ε, Ευρωπαϊκή ε, σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι συνέβη μετά το πραξικόπημα. και την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Ε, εκδόθηκαν, ε, αριθμός νομοθετικών διαταγμάτων. Στο πλαίσιο το συνταγματικό πλαίσιο η, ε, η κατάσταση της ανάγκης είναι αποδεκτή. Όμως, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν φαίνεται να συνάδουν με την συνταγματική τάξη. Για διάφορους λόγους. Πρώτον, λόγω της αρχής της αναλογικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 120 του συντάγματος, ε, το οποίο προβλέπει την κήρυξη κατάσταση έκτατη ανάγκη. Ο λόγο αυτή είναι η εξή. Είναι ε, η ύπαρξη βίων πράξεων που τείνουν να διασαλέψουν την δημοκρατία, να ανατρέψουν το δημοκρατικό καθεστώς. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι πολλά μέτρα είναι δυσανάλογα. Δεύτερον, έχουμε μέτρα που είναι ανσυνταγματικά. Τρίτον, μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. Τέταρτον, ε, μέτρα τα οποία είναι άσχετα με την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Πέμπτον, παραβίαση του δικαιώματο στην ιδιοκτησία, του δικαιώματο στην έκφραση και μέτρα τα οποία πλήττουν τον ε, βασικό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε οκτώ τύπους μέτρων που ε, δεν δικαιολογούνται από μια κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Είναι και αντισυνταγματικά και παραβιάζουν και την ίδια τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ε, η προθεσμία 30 ημερών κράτησης ε, είναι πολύ μακρά. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μέτρα τα οποία θα δώσουν αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα η διάλυση, το κλείσιμο νοσοκομείων, σχολείων κλπ. Δεν έχω χρόνο όμως να ε, δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό το θέμα. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι το εξής. Έχουμε σύνταγμα. Ένα σύνταγμα μεταμορφωμένο, διότι έχουν γίνει αναθεωρήσεις και μετατροποποίησεις από το 87 και μετά. Έχουμε όμως σύνταγμα. Αρκεί να το εφαρμόζουμε και να το σεβόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξομαλύνουμε ε, το συνταγματικό μας κράτος δικαίου. Όμως αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεκινήσουμε συζήτηση για μια νέα συνταγματική αναθεώρηση, διότι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε είναι εξαιρετικές. Για να γίνει σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν ήδη διατάξεις, δεν χρειάζονται καινούργιες, υπάρχουν ήδη διατάξεις αρκετές στο Σύνταγμα που θα μας επιτρέψουν να εξομαλύνουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έμα Σίγκλερ Βεπ έχει το λόγο τώρα. Human Rights Watch, Τουρκία, η Διευθύντρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μας προσκαλέσετε να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, όπως καταδικάζουν και συναδελφοί μου, το, την όπερα πραξικοπήματος του 15 Ιουλίου και την ε, απώλεια σε ζωές Καταδικάζω λίγο, ε, λοιπόν, και εγώ. Και για να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο ε, για τους θανάτους, ε, πήραμε συνεντεύξεις από άτομα στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, σχετικά με την απόπειρα βομβαρδισμού του Κοινοβουλίου, πώς απειλήθηκαν οι άμαχοι και όλα αυτά τα βάλαμε σε μια έκθεση. Πέρα από την απόπειρα πραξικοπηματός, θέλουμε να δούμε τι ακολούθησε, γιατί ο πληθυσμός της Τουρκίας υποστήριξε τη δημοκρατία εκείνο το βράδυ, απέτυσε τη δημοκρατία. Όμως, στη συνέχεια δεν τους δόθηκε η δημοκρατία, αλλά καταστολή και υπήρξαν επιπλοκές για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων εξαιτίας αυτών των ε, μέτρων. Δεν θα μπω σε νομική συζήτηση για την αναλογικότητα κτλ. γιατί το έχουν κάνει ήδη συνάδελφοί μου. Αλλά για να συνοψίσω, κάποια θέματα που αντιμετωπίσαμε μετά τα νομοθετικά ρητάγματα και την κήρυξη σε κατάσταση εκτακτού ανάγκης, Ε, ήταν ε, οι η δίωξη ατόμων συγγενικών ε, υποτιθέμενων υπόπτων που μπορεί να συμμετείχαν στο, στην απόπειρα 150 ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης έκλεισαν, έγιναν κατασχέσεις ιδιοκτησών κυρίως στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας και είναι μια κατάσταση όπου απλώ απλώς κατηγορεί κάποιον ότι είναι τρομοκράτη ώστε να χάσει την εργασία του στη δημόσια υπηρεσία ή να τον κλείσει στη φυλακή. Είναι πολύ, πολύ το κλίμα για τους πολίτες της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Με πάρα πολύ φόβο. Και η δυσκολία του να κάνουμε έρευνα είναι ότι πολύ λίγοι θέλουν να χρησιμοποιήσουμε τα ονόματά τους και αυτό θα οδηγήσει φυσικά στην ε, κατηγορία ότι τα δεδομένα που παρουσιάζουμε στην έρευνα δεν είναι αξιόπιστα γιατί δεν υπάρχουν ονόματα ούτε συγκεκριμένα. Γιατί έτσι δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν τις υποθέσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να εστιάσω στην εξαιρετική στο εξαιρετικό μνημόνιο μοράντουμ ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης που κάνει πολύ καλές συστάσεις σχετικά με τα νομιστικά διατάγματα και την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης παράλληλα αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιβολής ε, της ε, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης αρχικά 30 μέρες κράτηση. 5 μέρες χωρίς δικηγόρο. Όλα αυτά μας πάνε στο παρελθόν και είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονό αυτό, γιατί οι προηγούμενε ε, κυβερνήσει του AKP είχαν κάνει προσπάθειες προ τη βελτίωση. Γιατί το πρόβλημα που είχε η Τουρκία στο παρελθόν αντιμετωπίστηκε και βελτιώθηκε η κατάσταση από το ίδιο το AGP. Όμως με τέτοιου είδου μέτρα, τις συνθήκε κράτηση ανοίγουμε την πόρτα για μια οπισθοδρόμηση. Και αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη που δεν θα ήθελε η κυβέρνηση να συμβαίνει, γιατί αυτοί είχαν λάβει αυτά τα μεγάλα βήματα στο παρελθόν για να σταματήσουν τα βασανιστήρια. Κατηγορίε λοιπόν για βασανιστήρια κατά τη διάρκεια τη κράτηση κτλ. Είχαμε σχετικά με σχετικές μαρτυρίες ε, τις εβδομάδες ε, βασανιστήρια στρατιώτε που κρατήθηκαν εξαιτία του πραξικοπήματος. Φυσικά υπάρχει και θυμό ε, στι δυνάμει ασφαλεία, όταν αντιμετωπίζουν συνωμότε. Όμως θα πρέπει να μετριαστεί αυτός ο θυμός και από τις αρχές και από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε εξαιτία αυτού του φόβου, ε, αυτό το φόβο να κυριαρχήσει και τη διάρκεια της κράτη, το θυμό μάλλον, να υπερισχύσει. Συνεχίζονται να γίνονται πολύ σοβαρές ε, παραβιάσεις στην Οδό Βατάν, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Θα τα δημοσιοποιήσουμε όλα αυτά και θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυβέρνηση γιατί να γνωρίζουμε ότι προφανώς δεν θα θελήσουν να συνεχιστούν όλα αυτά και θα θελήσουν να λάβουν κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ακόμα δύο σημεία που θέλω να θίξω. Το, η έκθεση του ε, CPT θα θέλαμε να εκδοθεί. Θα ήταν πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση γιατί θα υποφελούνταν από ε, τα πορίσματα αυτή τη έρευνα. Αλλά είναι στη κριτική ευχαίρεια της κυβέρνηση, αν θα δημοσιοποιηθεί ή όχι πρόθεσμα. Είμαστε απογοητευμένοι που ο ειδικό συζητητή για τα βασανιστήρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Χουάν Μέντε, δεν του επιτράπει είσοδο στην Τουρκία για να ερευνήσει τι ε, ε, συνθήκε κράτηση. Ε, όταν θα του επιτραπεί, θα είναι μάλλον κάποιος νέος ε, εισηγητής. Πρέπει να γίνει όμως αυτό χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει να υπάρξει επιτήρηση στα σημεία κράτηση, να γίνουν ad hoc επισκέψει σε σημεία κράτηση και σε φυλακέ, ακόμα και για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το θέμα της κράτηση είναι μια μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή και η Τουρκία δεν θέλει να ισχύει αυτό, δεν θέλει να το βλέπουμε έτσι το θέμα. Θα περάσω στην ενοχοποίηση ατόμων για τη συμμετοχή σε οργανώσεις. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα σε σχέση με, με, το, με τη συμμετοχή στο ΠΚΚ. Συμμετέχουν στο ΠΚΚ, ανεγραμμένοι γεγραμμένοι ότι είναι τρομοκράτες. Το ίδιο ισχύει και τώρα, καθώς η κυβέρνηση διατείνεται ότι οι οπαδοί του Φετουλάχ συνιστούν τρομοκρατική οργάνωση, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πολλοί άνθρωποι όπως δάσκαλοι και τα λοιπά, οι οποίοι υποστηρίζουν τις ιδέες του Φετουλάχ Γκιουλέν, θεωρήθηκαν τρομοκράτες. Αυτή είναι μια προσέγγιση που δεν είναι έγκυρη, γιατί θα πρέπει να βασίζεται σε εγκληματικές πράξεις αυτός ο χαρακτηρισμός. Και αυτό δεν ισχύει προς το παρόν. Έχει απλωθεί ένα δίχτυ ενοχής. για άτομα που είναι σε επικοινωνία με το Τσιμπάτ και άλλες οργανώσεις. Γιατί αυτό αφορά την μισή, τον πληθυσμό της Τουρκίας. Με τον άνθρωπο με τον άλλον είναι σε επαφή με γκυλενιστές. Είναι όλοι αυτοί επομένω τρομοκράτες. Είναι πολύ προβληματική αυτή η προσέγγιση. Ελπίζουμε όλα αυτά το γρήγορα να μετριαστεί. Πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι πολλοί εισαγγελείς και δικαστές ε, είναι στη φυλακή. Έχω νούμερα, 34.000 ε, προκρατούνται, 77.000 θα οδηγηθούν σε δίκη. Είναι τεράστια τα νούμερα, 2.300 δικαστές θέλουν υποκράτηση, υπάρχει έλλειψη στοιχείων για την κράτησή του, είναι λυπή τα στοιχεία για την κράτησή του σύμφωνα με αυτά που έχουμε εξετάσει μέχρι στιγμή. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο, ελευθερία του τύπου, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Η καταστολή της ειρηνευτικής διαδικασίας ε, στα νοτιοανατολικά. πάνω στην οποία αναπόθεσαν πολλέ ελπίδε ε, οι Κούρδοι και όχι μόνο, ολόκληρο ο πληθυσμό τη Τουρκία που θέλουν άμεσα στο μέλλον να σταματήσει αυτή η διαμάχη. Η κατάσταση του τελευταίου μήνε. οδήγησε στον εκτοπισμό 400.000 ατόμων από τα νοτιοανατολικά όπου υπήρξαν σειράξει στα κέντρα των πόλεων, τεράστιες καταστροφές όπου γίνεται και κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλε τι πλευρέ που συμμετέχουν στην ε, διαμάχη στη σύραξη αυτή. Άλλο ένα θέμα που δεν έχει να κάνει άμεσα με το πραξικόπημα, αλλά που δείχνει ότι κάποια μέτρα αποτέλεσαν ε, κατασταλτικά, ε, ε, λειτουργήσε κατασταλτικά σε μέσα με ενημέρωσης της κουρδικής πλευράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, έχει το λόγο η κυρία Σιμών Γκαμποριό, λέει πρόεδρος, από το Μεντέλ, Ευρωπαϊκή Δικαστική για την Ελευθερία Θα έχουμε και λίγο χρόνο για να τοποθετηθείτε και οι υπόλοιποι βουλευτέ. Το δεκάμιση πρέπει να φύγουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σα. Σα μιλάει ένα δικαστή με πρόεδρο του στο επίτιμη, στο εφετείο του Παρισιού και ιδρυτικό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, Δικαστών για τη Δημοκρατία και τι Ελευθερίε. Θα σα μιλήσω εξ ονόματος μιας πλατφόρμας όλων των οργανώσεων Ευρωπαίων δικαστών που έχει συγκροτηθεί ένα ιστορικό γεγονός γιατί ποτέ δεν ήμασταν ενωμένοι. Για ποιο λόγο. Είναι αυπρεγουμένο αυτό το γεγονός. Αυτή τη στιγμή 2.845 δικαστές βρίσκονται σε κράτηση. Κρατούνται με την επιφύλαξη κάποιου φάρματος γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. 3.390 ανακλήθηκαν από τις θέσεις τους λόγω συλλογικών, συλλογικών διαταγμάτων, για ανάκληση των θέσεων τους. Υπήρχε κατάλογος με ονόματα στην επίσημη εφημερίδα 3.390 που απομακρύθηκαν από τις θέσεις τους. Αυτοί οι δικαστές δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Όλες οι περιουσίες τους δημεύτηκαν Τα ονόματά τους δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα και διαπομπεύθηκαν. Πώς μπορούν να βρουν εργασία τη στιγμή που τους αποκλείεται, απαγορεύεται η πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικαστικό επάγγελμα και θεωρούνται από, το, από την κοινή γνώμη ως τρομοκράτες. Δεν βρίσκονται, δεν είναι περάνω του νόμου οι δικαστικοί. Βεβαίως και μπορούν να διωχτούν πειθαρχικά ή ποινικά, αλλά βάσει δίκαιων διαδικασιών όπου έχουν το δικαίωμα έκφρασης και όπου τα αποδεικτικά στοιχεία τους κοινοποιούνται. Οι δικαστές έχουν δικαίωμα, όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι. Και πέραν των δεινών που αντιπροσωπεύει αυτούς και τις οικογένειές τους η φυλάκηση υπάρχουν υψηλότερες αξίες που αμφισβητούνται γιατί ο κάθε δικαστικός είναι ένα μικρό κομμάτι της δικαστικής εξουσίας που εκπροσωπεί. Τι να σας πω τώρα βέβαια σε πέντε λεπτά είναι αδύνατο να σας περιγράψω τα πράγματα πλήρως. Να σας πω όμως καταρχάς ότι ήδη εδώ και πολλά χρόνια εμείς ενός ευρωπαϊκού Ευρωπαίων Δικαστών λέμε συνεχώς ότι προσοχή το κράτος δικαίου στην Τουρκία που ήδη είχε κάνει αρκετά βήματα πρόοδου απειλείται ήδη από την άνοιξη του 2015 είχαν φυλακιστεί έξι δικαστές επειδή ακριβώς είχαν ασκήσει διώξεις ή είχαν αφήσει ελεύθερα κάποια άτομα και ακόμα δεν έχουν δικαστεί. Κρατούνται ακόμα εδώ και 18 μήνες ενώ οι δίκες τους καθυστερούν πολύ. Δικαστές επίσης μετατοπίστηκαν με τρόπο μάλλον αυθαίρετο, περισσότερο παρά λιγότερο αυθαίρετο. Πήγαν από το στον νότο της χώρας, κοντά στα σύνορα με την ε, Συρία, επειδή έλαβαν αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν αρεστές στους ανωτέρους τους. Σιγά σιγά σιγά είχαμε λοιπόν μια υποβάθμιση της δικαστικής εξουσίας και της ανεξαρτησίας της. Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης που εξελέγει το 2014 εξελέγει υπό συνθήκες πολύ ύποπτες. Υπήρξαν πιέσεις προς τους δικαστές και μία νέα οργάνωση δικαστών συγκροτήθηκε κοντά στην εξουσία και αυτοί ακριβώς κατέλαβαν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και αυτοί συνέβαλαν βεβαίω σε αποφάσεις οι οποίες είναι τελείως αμφισβητήσιμε όπως η απομάκρυση των δικαστικών από τους. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι να γνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να κρατήσει άλλο. Θα ήθελα να παραθέσω τον υπαταρμοστή ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν είπε ότι αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την Τουρκία να, να αποδείξει ότι ακόμα και σε, ένα, σε περιστάσεις όπου 300, 300 δικαστές ε, απομακρύνθηκαν τις θέσεις τους και φυλακίστηκαν, το πώς τα τουρκικά δικαστήρια θα μπορέσουν να αποτρέψουν τι ενδεχόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω ακριβώς το αυθαιρέτων αποφάσεων του εκτελεστικού ή της διοίκησης ή ακόμα και την ίδια τη δικαστική εξουσία. Επειδή ακριβώς αυτοί οι δικαστές απομακρύθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους τους και διώκονται από τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Θα πρέπει να απογραμμίσουμε λοιπόν ότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει προσφυγή κατά αυτών των μέτρων γιατί έχουν χαρακτήρα νόμου. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την υπόθεση. Πάντως, στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή 20.000 προσφυγές μετά από τις αντιδράσεις που είχαμε μετά το πραξικόπημα. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν έχουμε μια ε, διεκδίκηση συντεχνιακή. Απλά και μόνο πρέπει να πούμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι πια αδίκαστη, δεν είναι πια ανεξάρτητη, είναι πια αδύνατο να έχει κανείς στην Τουρκία εφαρμογή δικαίου με τρόπο δίκαιο. Αυτοί οι δικαστές δεν είναι απλά ονόματα ή απλοί αριθμοί ή κάτι το, το αφηρημένο. Τους γνωρίζω προσωπικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας νάλφος που είχε έρθει στη Γαλλία πέρσι για να, να μας δώσει τη μαρτυρία του για την κατάσταση είναι φυλακισμένος. Κρατείται σε ένα κελί που προβλέπεται για 9 και είναι 32 μέσα. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κίνδυνος, σοβαρός κίνδυνος συγκεκριμένη συμπεριφοράς, επιθετικής, όταν ε, κρατείται κάποιος σε σε τέτοιες συνθήκες υπάρχουν και υπάρχει το ενδεχόμενο επιθετική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δέχονται λοιπόν πιέσεις, εκφοβισμούς, και μάλιστα ο ίδιος ο ο εκπρόσωπο των δικαστικών στην Τουρκία έλαβε θέση κατά των συναδέλφων του. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τους ε, βοηθήσουμε αφιλοκερδός. Αλλά μια κόρη ενός δικαστικού που γνωρίζω μου είπε ότι ο πατέρας μου δεν θέλει να δεχτεί βοήθεια από έναν ξένο δικαστή. Γιατί δεν θα το επιτρέψουν να έχει δικαίωμα προσφυγή. Δεν επιτρέπουν σε τουρκου δημοσιο... ε, να του βοηθήσουν. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση βρισκόμαστε και εξ ονόματο αυτή τη πλατφόρμα. θα μπορούσα βέβαια να σα είχα και ένα λεπτομερέστερο κείμενο με πολλά που θα είχαμε να πούμε, αλλά εντάξει δεν έχουμε χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε αυτά τα λίγα που σα είπα δεν είναι καν αντιπροσωπευτικά του μεγέθου τη κατάσταση Πάντως εμείς θρηνήσαμε τα θύματα του πραξικοπήματος, αλλά θρηνούμε και τα τωρινά θύματα αυτής της αυθαίρετης καταστολής. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Είχαμε το 2010 όταν έκανε σοβαρές μεταρρυθμίσεις ώστε η τουρκική δικαιοσύνη να γίνει ουσιώδης, ε, αδίκαστη, ανεξάρτητη. Και το Σταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας έλαβε υποδειγματικές και θαραλές αποφάσεις. Θα πρέπει οι δικαστές λοιπόν να είναι ανεξάρτητοι. Αν λοιπόν δέχονται πλήγματα από πολιτικούς στην Τουρκία, δεν είναι ότι υπήρχαν κάποια σχέση με τον Κιουλέν, απλά και μόνο επειδή έκαναν το καθήκον τους. Και εμείς εδώ κάνουμε και λαμβάνουμε αποφάσεις στην Γαλλία κατά πολιτικών και δημοσίων ε, προσώπων. Σε όλες τις χώρες γίνεται αυτό. Δεν, σημαίνει ότι θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από τις θέσεις μας. Δυστυχώς, λοιπόν θρυνούμε, θρυνούμε γιατί χάνουμε όλο και περισσότερο αυτή την εμπιστοσύνη την οποία θα θέλαμε να ανακτήσουμε. Θέλουμε λοιπόν να ε, είμαστε σε θέση να εμπιστευόμαστε την, την Τουρκία ώστε να μπορέσει ακριβώς να θεσπίσει ένα κράτος δικαίου άξιο αυτού του μεγάλου λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, όλους τους ε, ομιλητές. Θα δώσω το λόγο τώρα την Προεδρία μάλλον στον κύριο Κεφαλογιάννη που είναι και συμπρόεδρος. Ε, θα δίνει το λόγο στους διάφορους συναδέλφους. Ε, μέχρι τις μία παρατέταρτο έχουμε πλέον χρόνο. Καταφέραμε και πήραμε μία παράταση έτσι ώστε να πάρετε και εσείς το λόγο και να απαντήσουν οι ομιλητές μας. Ο λόγο τώρα στα μέλη μα, Ο κ. Γκίλ καταρχήν. Γκίπ, συγγνώμη. Ο κ. Γκίπ. Δεν κατάφερα να πάρω το λόγο στο πρώτο κομμάτι της συνάντησης που μας μίλησε ο ε, Υφυπουργό. Ε, είχαμε πολύ λίγο χρόνο και τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Δεν καταφέραμε να ε, θέσουμε ερωτήσει όλοι μας, αλλά η ερώτηση εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη μα έκανε μια εξαιρετική έκθεση για την εσωτερική κατάσταση. Και νομίζω όλοι μετά υπογράμμισαν ορισμένα πράγματα. όλοι είπαμε ότι είμαστε αντίθετοι με το πραξικόπημα η συνταγματική τάξη δεν μπορεί να διακοπεί από πραξικοπήματα. Δεν μπορεί να διακόπτεται από πραξικοπήματα. Όμως ε, η, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να βοηθηθεί η Τουρκία για να διατηρήσει το κράτος δικαίου. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ωφέλιμο για όλους. Η Τουρκία θα πρέπει να επιστρέψει και στη διεθνή σκηνή ισχυρότερη. Επίσης, πώς βλέπετε τη θανατική ποινή ε, σε σχέση με τα γεγονότα αυτά. Ε, θα πρέπει να όλοι μας επιθυμούμε η Τουρκία να είναι μια σταθερή χώρα, ετερός. Αξιόπιστο εταίρος τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μια χώρα με την οποία μπορούμε να διατηρούμε καλές σχέσεις. Και αυτό λόγο γίνεται και η σημερινή ακρόαση, για να ακούσουμε την άποψη τόσο τη κυβέρνηση όσο και άλλων παραγόντων και διεθνών οργανισμών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάτι Πύρη είναι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Αμέσως μετά το πραξικόπημα ε, δημιουργήθηκε μια ευκαιρία για την Τουρκία. Πολιτική ενότητα, ομοψυχία, χρειαζ... Ε, ε, φάνηκε ότι χρειάζεται πολυφωνία. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να προστατεύσει την δημοκρατία και η Τουρκία είχε διεθνή στήριξη. Δύο μήνες μετά δυστυχώς βλέπουμε ότι ε, έχει παρατεθεί η κατάσταση εκτής, ε, ε, κατάστασης, ε, χιλιάδες συλλήψεις ε, κλπ. Ερώτηση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχετε δημιουργήσει ή δημιουργείται ένα σύστημα παρακολούθησης κατάσταση. Συμφωνώ με τα όσα είπαν ορισμένοι ομιλητέ ότι είναι πολύ σημαντικό η τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει τη δημοσίευση τη έκθεσης της Επιτροπής ε, πρόληψη Βασανιστήριων. Επίση, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν λαμβάνουν χώρα βασανιστήρια. Αυτό είναι ο τρόπο να αντιμετωπιστούν οποιασδήποτε καταγγελίε. Επίση, Έμα, Έμα Σενκλέρ, ε, ανέφερε στην κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αυτή τη βδομάδα βλέπουμε ακόμα περισσότερη κλιμάκωση τη διαδικασία Το ΠΚΚ δολοφονεί υψηλά στελέχη του κόμματο δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να στρέψουμε και εκεί το βλέμμα μα στην κλιμάκωση στην νοτιοανατολική Τουρκία. Τελευταία ερώτηση για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που βρίσκονται εδώ. Ε, συζητάτε και με Τούρκους βουλευτές και με την τουρκική κυβέρνηση στην Τουρκία ή εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μόνη θέση, ο μόνος τόπος στον οποίο έρχεστε σε διάλογο με την τουρκική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κυρία Ροντρίγκε, θα μιλήσω στα Πορτογαλικά. Ε, Επισκέφθηκα την ε, Τουρκία με αυτή την επιτροπή δύο μήνες πριν την απόπειρα πραξικοπήματος. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πιο, το πιο κατάλληλο φόρουμ για να συζητήσουμε ειλικρινά όλα αυτά τα θέματα. Με διαφάνεια όμως. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές, ιδιαίτερα τον κύριο Κορκού, τον οποίο είχα συναντήσει. και Είχαμε πάρει πρωινό μαζί και στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα όμως να πω κάτι άλλο και θα μιλήσω αργά-αργά για να με καταλάβετε. Ποιο αποφάσισε αυτό το πραξικόπημα. Όταν εμείς πήγαμε στην Τουρκία, ήμασταν τρει ευρωβουλευτέ, ε, μας ε, τέθησαν στην υπόψη μας διάφορα θέματα. Τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωση για την ένταξη Τουρκίας, οι οργανώσεις με τις οποίες συναντηθήκαμε όλε Μα είπαν ότι υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα, ε, απόκληση μάλλον ανάμεσα στο Σύνταγμα και τους νόμους της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα τις ε, ε, αποφάσεις ε, σύλληψης, ε, ε, το κλείσιμο διαφόρων sites στο ίντερνετ και περιορισμού στην πρόσβαση, διώξη εναντίον ακαδημαϊκών, χειραγωγής της δικαιοσύνης, χρηματοδότηση μόνο οργανώσεων που στηρίζουν την κυβέρνηση, φιλοκυβερνητικών οργανώσεων, η ελευθερία έκφρασης, το θέμα των προσφύγων και εκεί θα πρέπει να πω ότι η Τουρκία είναι πολύ γενναιόδορη. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζονται δύο μηχανισμοί ε, λογοδοσίας και εσωτερικός και εξωτερικός προκειμένου να προσπιστούν οι ζωές τους. Τώρα, το κράτος, η κατάσταση έκτατης ανάγκης. Ε, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια περίπτωση αναστολής του δικαίου. Αναστολής του κράτους δικαίου. Ε, αυτή η αναστολή του κράτους δικαίου ε, δεν μπορεί να οδηγεί σε κατάχρηση της από το κράτος. Το βράδυ της 15ης Ιουλίου ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους για να προστατεύσει τη δημοκρατία του. Μια και έχουμε εδώ εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, άργησε μάλλον να τοποθετηθεί έναν του πραξιοπήματος. Την επόμενη μέρα είπα ότι η εκπρόσωπος για τις εξωτερικές μας σχέσεις ε, τοποθετήθηκε ακριβώς την επόμενη μέρα. Πάνω από 200 νεκροί βέβαια, αλλά πάνω, ε, περισσότερο 50% αυτών ήταν μεταξύ των πραξικοπηματιών. Έτσι να διορθώσω και αυτό. Συγγνώμη, έχουμε 16 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό το πραξικόπημα στην Τουρκία. Αυτό είναι, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, εισηγητές, πολύ σημαντικέ οι πληροφορίε που μας έδωσαν. Θέλω να αυτό που είπε η κυρία Καμπόριου, ναι, κλαίγαμε με τους ανθρώπους της ε, Τουρκίας ε, το βράδυ του παραξικοπήματος και τώρα και με αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή και που διώκονται αδίκως. Η ερώτησή μου είναι τι θα κάνουμε μετά, γιατί ήμασταν καλοί στο να δείξουμε ε, τη συμπαράσταση καταδικάζοντας ε, το... το πραξικόπημα αλλά και τις αρχές και θα πρέπει όμως από εδώ και πέρα να εμπλακούμε σε ένα διάλογο για το μέλλον γιατί αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος είναι να υποστηρίξουμε την Τουρκία, τον λαό, όχι την κυβέρνηση, τον λαό της Τουρκίας για να ε, προχωρήσει σε μια μακροπρόθεσμη δημοκρατική μεταρρύθμιση που να ε, ε, συμπεριλαμβάνει όλες τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ ξεκάθαρος. Μπορεί να είστε ξεκάθαροι, σαφείς στις διατυπώσεις και να μας πείτε επίσης τι γίνεται στις φυλακές, στα κέντρα κράτησης, που έχει σχέση με αυτό που είπε η κυρία Σενκλέρ. Είναι το πιο ανησυχητικό θέμα αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να απασχολεί την κυβέρνηση της Τουρκίας και που πρέπει να το αλλάξει. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις αρχές της Τουρκίας και τους φιλελεύθερους που μας λένε ότι η Ευρώπη μας γυρίζει την πλάτη γιατί δεν αναγνωρίζεται ότι το τραύμα του προεξοπήματος είναι για όλη την κοινωνία. Και όπως είπατε κύριε Κόρκ, αυτό που είναι κατανοητό ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι πρέπει να εργαστούν. Πώς μπορούμε να ε, κάνουμε τη διαφοροποίηση, τη διαφορά για αυτούς που, ε, ε, διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το πραξικόπημα και αυτούς που υποστηρίζουν τον Γιουλάχ και δεν ευθύνονται για το πραξικόπημα. Πώς μπορούμε να είμαστε υποδομητικοί και να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα ώστε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις του μέλλοντος. Η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Αυτό που είπε η κυρία Καμποριέου. Η πρόσβαση στις φυλακές είναι απαραίτητη. Η Τουρκία, αν υπάρχει αυτοσεβασμός στην κυβέρνηση, θα πρέπει να επιτρέψει τους συγκητές των ΗΠΑ και αποστολές ε, λεφτών να μπουν στις φυλακές και να ελέγξουν την κατάσταση σχέση με τα βασανιστήρια και με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρουλάκη παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου μιλητή. Όποιος διαβάζει τι σημαίνει στην Τουρκία κατανοεί ότι το κράτος δικαίου επλήρεται βάναυσα ότι υπάρχει καθημερινή παραβίαση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και είναι παράλογο να θεωρούμε ότι όλα αυτά ξεκινούν στις 15 του Ιούλη. Δηλαδή ήρθε ο υπουργό, έκανε εδώ μία ανάλυση και μας είπε ότι μετά τις 15 Ιούλη που κανείς από εμά προφανές δεν ήθελε η Κούντα να έχει μια δικτατορία, στηρίξαμε με κάθε τρόπο τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, ότι μετά τις 15 Ιούλη ξεκινούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία εμείς καταδικάζουμε ή μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο ω παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Διότι ο τρομονόμο ο οποίο οδηγούσε σε άρση ασυλία βουλευτών Κούρδων έγινε πριν τι 15 Ιουλίου. Στις τηλεοράσει μας βλέπαμε στα μέσα μαζική ενημέρωση, ότι το κλείσιμο εφημερίδων και η φυλάξη δημοσιογράφων συνέβαινε και πριν τι 15 Ιουλίου. Και αυτό που θέλω από εσά είναι να μα πείτε τελικά τι ήταν αυτό που οδήγησε στο πραξικόπημα τη Τουρκία και σε όλη αυτή την κατάσταση. Και δεύτερο, τι πρέπει να κάνει, τι προτείνεται ότι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να στηρίξει τα συμφέροντα του τουρκικού λαού που είναι καθαρά να υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα ισχυρό κράτο δικαίου ώστε να υπάρχει ευημερία και προοπτική ευρωπαϊκή για το λαό του τουρκικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δουλάκη. Ε, ε, ευχαριστώ. συμφωνώ ότι τα πράγματα δεν ξεκίνησαν την 15η Ιουλίου. Αν ακολουθήσουμε τις ε, ομάδες, τα κόμματα και τους, ε, τις δηλώσεις και των ομάδων και των ε, ευρωβουλευτών, την αυξανόμενη ανησυχία μας για την χειροτέρευση της κατάστασης στην Τουρκία. Δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος Ερντογκάν οδηγεί τη χώρα σε μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Πρόεδρος. Αλλά όπως υπόθηκε και πριν, καταδικάζουμε πλήρως την απόπειρα πραξικοπήματος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις δυνάμεις που κρύβονται πίσω από αυτό. Έχουμε μια εξαιρετική έκθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Επιτρόπος έκανε εξαιρετική δουλειά ένα δέκα σελίδων έγγραφο το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους μας. Θέλω να ρωτήσω τους εισηγητές κατά, κατά πόσο συζητείται αυτό το έγγραφο στην Τουρκία μεταξύ πυρογνωμόνων. Γιατί από την πρώτη σελίδα υπάρχουν όλες οι προτάσεις και οι συστάσεις. Αν τις εφαρμόσετε, τα πράγματα θα καλυτερεύσουν πολύ γρήγορα. Κατά πώ θα αξιοποιείται αυτό το έγγραφο στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Σε 7 λεπτά, λέει ο Πρόεδρο, θα σταματήσει η διερμηνία. Μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά, αλλά θα σα παρακαλούσα να ε, κάνετε τη δήλωσή σας ε, μέσα σε ένα λεπτό. Κύριε Μαυρίτη, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο, Ένα λεπτό. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι η συστηματική παραβίωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα θέμα βαθμού στην Τουρκία. Όσον αφορά το θέμα μας, Τουρκία και το κράτος δικαίου. Δεν θα μιλήσω για τους ακαδημαϊκούς, τους δασκάλους, τους δημοσιογράφους. Θα επικεντρωθώ στο δικαστικό σύστημα. Χιλιάδες είναι στη φυλακή ή στιγματισμένοι. Και αυτοί προέρχονται από το δικαστικό σώμα. Η επόμενη ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Από ευρωπαϊκή σκοπιά και πρέπει να τολμάμε να θέτουμε αυτό το ερώτημα. Μπορούμε να έχουμε κράτος δικαίου, να έχουμε μια δημοκρατική κοινωνία σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Και θέλω μια απάντηση σε αυτό. Κυρία Βέργια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επανέλθω σε αυτό που είπαν πολλοί συναδελφοί. Και εγώ εξεπλάγιν ακούγοντα τον Υπουργό που έλεγε ότι δεν είχαμε καταδίκες από την Ένωση. Νομίζω όλοι καταδικάσαμε την απόπειρα πραξικοπήματος και μάλιστα μας εξέπληξε η πορεία της κατάστασης στη συνέχεια και είμαστε πολλοί που διαπιστώσαμε ότι είχαν υπάρξει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια όσον αφορά ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Αλλά όπως υπόθηκε εδώ και πολλά χρόνια τα πράγματα επιδεινώνονται. Και μάλιστα είχαμε την εντύπωση κάποιοι παρατηρητές ότι ήταν πρόσχημα η απόπειρα για την επιδείνωση της κατάστασης. Και βέβαια αυτό είναι δραματικό σε σχέση με την εξέλιξη της κατάστασης. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, κυρίως την κυρία Σανκλέρ, που επέστησε την προσοχή μας για αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Τουρκία. Γιατί πράγματι αυτά δεν εξισώνονται. Ο ορισμός τρομοκρατικής οργάνωσης είναι ένα θέμα κλειδί. Το είπε όμως πολύ καλά ο προηγούμενος ομιλητής. Είναι το σημείο κλειδί του, δικαστου, του δικαστικού συστήματο και το τι σημαίνει με του δικαστέ. Έτσι και κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ για ελευθερία έκφραση το πρωί. Νομίζω αυτό είναι θεμελιώδε και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιε ανασταλές λειτουργία τηλεκμιακών οργανισμών λόγω ακριβώ τη απόφαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κ. επιτήριο για ένα λεπτό, ο κ. Λόπε και μετά θα δώσω το, το λόγο δύο λεπτά στον Υφυπουργό και δύο λεπτά σε ε, τους πανελίστες. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Λαμπέ, ναι, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει συστηματική παραβίαση του χαμπέας κόρπους στην Τουρκία, βασικό θεμελιώδε στοιχείο του κράτους ε, δικαίου που επιτρέπει ακριβώς την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και την δικαστική ευθερεσία. Αυτό παραβιάζεται συστηματικά στη χώρα. Και εμείς αυτό το λέμε εμείς ξεκάθαρα, έχοντας καταδικάσει ενεργά την απόπειρα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Να προσθέσω κάποια πράγματα σε σχέση με τις δημεύσεις και εθνικοποιήσεις ε, κάποιων επιχειρήσεων. Βεβαίω δεν είναι το ίδιο ως παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, αλλά βεβαίω και αυτό έχει επιπτώσει στην δικαστική ασφάλεια. Και μετά με, τα βασανιστήρια, τι γίνεται, έχουμε βασανιστήρια στι φυλακέ τη Τουρκία. Και τελευταίο ερώτημα. Αφού εξετάζουμε την κατάσταση πέραν της απόπειρας, πραξικοπήματος, αυτό που βλέπουμε είναι μια αλλαγή στην ταυτότητα και στην φύση του τουρκικού κράτους. Δηλαδή μια ρήξη με, τα, με τις ιδρυτικές αρχές της σύγχρονης Τουρκίας που έχουν να κάνουν με το κράτος ε, δικαίου και τη σχέση της χώρας αυτής με την περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Σοπιτίδιος. Πρόεδρε, πολύ σύντομα θέλω να ρωτήσω με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην τουρκική δικαιοσύνη πώς είναι δυνατόν να υπάρξει αμεροληψία μεταξύ των δικαστών οι οποίοι διώκονται κατά τον τρόπο που διώκονται. Πώς είναι δυνατόν να διεξαγάγουν δίκαιες δίκες όταν επάνω από το κεφάλι τους επικρέμαται η δαμόκλειο σπάθη του καθεστώτος της Τουρκίας. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να αποδείξει την αθωότητά του. Τι στη μαρτυρία θα επικαλεστεί ότι δεν είναι μέλος τρομοκρατικής οργανώσεως και τι θα απαντήσει στο ερώτημα και πού ξέρει εσύ εάν όχι είναι μέλο τρομοκρατική οργανώσεω. Ήσουν εσύ μέλος τη της οργανώσεως, ώστε να μην τον δει εκεί. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και είναι πολύ δικαιολογημένη η ανησυχία και τα ερωτήματα που θέλετε για βασανιστήρια, για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. όμω εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, επειδή γνωρίζουμε ποια είναι η Τουρκία και πώ λειτουργεί, ότι θα ισχύσει αυτό που είχε πει ο Βρένο. ουέ τη ιτημένης. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Κυρία τελευταία μιλήτρια. Α, όχι, πρώτη τελευταία. Το κύριο Σελήν. Ο κύριο Σαχίν. Α, ο υφυπουργό. Ο κύριο Σαχίν, παρακαλώ, δύο λεπτά. Σέβομαι όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν. Ακούω και τις επικρίσεις. Εδώ στις Βρυξέλλες αισθάνομαι Υπάρχει μετάφραση, υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, βλέποντας τα πράγματα από εδώ και ακούγοντας τις επικρίσεις φαίνεται σαν να κάναμε λάθος που ε, αντισταθήκαμε στο πραξικόπημα στην Τουρκία. Ε, αυτό που ζήσαμε ήταν μια προσπάθεια διασάλευσης της ε, συνταγματικής τάξης. Ήταν μια προσπάθεια περιορισμού των δικαιωμάτων. Οι ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άνθρωποι τραυματίστηκαν, βομβαρδίστηκαν κρατικά κτίρια, ε, το προεδρικό μέγαρο. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Και τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να τα κατακρίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μην ξεχαράμε το εξής. Πριν από τρία χρόνια, στην Τουρκία, ε, έγινε η δίκη ε, ε, εργενεκών, του σκανδάλου εργενεκών και είδαμε ότι τελικά ε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταδικαστεί βρήκαν το δίκιο τους και αθώθηκαν. Αυτό αποδεικνύει την ανεξαρτησία της Η αθώωση αυτών των ανθρώπων το αποδεικνύει. Η κατάσταση εκτεκτής ανάγκης και τα αντίστοιχα νομοθετικά διατάγματα εγκρίνονται από τη Βουλή. Δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως και υποστηρίζονται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Η Βουλή, επαναλαμβάνω, έχει δικαίωμα να απορρίψει ή να τροποποιήσει αυτά τα νομοθετικά διατάγματα. Ασφαλώς θα πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονική συνταγματική τάξη το συντομότερο. Και από πλευρά εσωτερικό και από πλευρά διεθνού δικαίου. Τελευταία μου κουβέντα. Μία φράση ακόμα. Σε ό,τι αφορά, τα, ε, σε την Human Rights Watch και την εκπρόσωπη. Ε, δεν αναφέρθηκε καθόλου στις ε, σε στελεχών του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δεν αναφέρθηκε καθόλου στη βομβαρδισμό ε, κρατικών κτίριων από τρομοκρατικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς και συνεχίζουμε στα αγγλικά και τα γαλλικά. Mrs.